Uh, Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Ας περάσουμε στο επόμενο σημείο της σημερινής ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής ΑΦΕΤ, που είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Εξωτερικών Υποθέσεων της Δημοκρατίας της Παραγουάη και που είναι υπεύθυνο και έχει αναλάβει προσωρινά την Προεδρία της Μερκοσούρ. Καλώς ήρθατε λοιπόν κύριε Αντώνιο Ρίβας είναι μαζί μας, όπως είπα και πριν, για να εκπροσωπήσει τη Μερκοσούρ, που αποτελείται από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Ορουάη και την Παραγουάη. Είναι μια πάρα πολύ καλή στιγμή λοιπόν που σας έχουμε εδώ μαζί μας ε, σήμερα, γιατί οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Μερκοσούρ βρίσκονται ψηλά ψηλά στην ημερήσια διάταξη. Στις 28 Ιουνίου του 2019, μετά από 20 χρόνια διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μερκοσούρ κατέληξαν σε συμφωνία επί της αρχής για τον εμπορικό πυλώνα ε, στα πλαίσια μιας ευρύτερης συμφωνίας σύνδεσης που περιλαμβάνει πολιτικό διάλογο και συνεργασία. Η συμφωνία αυτή περνάει από νομική αναθεώρηση πριν ε, μεταφραστεί και υποβληθεί προς ε, επικύρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μερκοσούρου θα μπορούσε να έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία ιστορική θα έλεγα και για τις δύο περιοχές ε, του κόσμου, όχι μόνο οικονομικά αλλά και πολιτικά. Εφόσον επικυρωθεί θα δημιουργούσε την μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με την οποία, την οποία έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα καλύπτει πληθυσμό πάνω από 780 εκατομμύρια και θα επαγιώσει ακόμα περισσότερο τις στενές πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές ε, σχέσεις και δεσμούς μεταξύ των δύο περιοχών. Σήμερα με τη Μερκοσούρ δείχνουμε ότι εμείς θέλουμε να διατηρήσουμε την διεθνή τάξη που να βασίζεται σε κανόνες μέσα σε μια στιγμή πολλών ε, προκλήσεων και με πολλούς ε, παίχτες που βρίσκουν το δρόμο τους ε, στο πολυμερές επίπεδο. Έχουμε δεσμευτεί λοιπόν να προωθήσουμε τη διεθνή συνεργασία για θέματα όπως είναι η κλιματική αλλαγή, το εμπόριο, η διεθνή συμφωνία κτλ. Όλα αυτά επηρεάζουν και άλλα ζητήματα που πρέπει να κοιτάξουμε, ανθρώπινα δικαιώματα κλπ. Προσβλέπουμε λοιπόν στη συζήτηση μαζί σας για να μάθουμε ποια είναι η κατάσταση πραγμάτων κατά τη γνώμη σα για τη σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση και Μερκοσούρ. Προηγουμένω όμω, θα δώσω το λόγο στον Νίκολα Ντάντι που είναι ο πρώτο αντιπρόεδρο τη αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι σχέσει μα με τι χώρε Μερκοσούρ. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, να χαιρετήσω τον Πρωθυπουργό για την παρουσία του, τον Υπουργό εδώ για την παρουσία του. Είχαμε ειδωθεί στην Ασουνθιόν όταν πριν από λίγου μήνε είχαμε πάει εκεί με την αποστολή τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την παρακοτήρηση των ε, εκλογών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια συνεργάζεται με την Παραγουάη, διότι μας έχει ζητηθεί υποστήριξη κατά τη διάρκεια των εκλογών και το 2016 και το 2018. Και επ' αυτού, Υπουργέ, περιμένουμε τους ερχόμενους μήνες και εβδομάδες η Παραγουάη και η Βουλή της χώρας να αποστείλει σημαντικά μηνύματα για να προωθηθούν κάποια σημεία που είχε τονίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα πρέπει να προωθηθούν. Στην τελική μας έκθεση του 2018 έχουμε πολλά προγράμματα συνεργασίας σημαντικά μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Παραγουάης και σας ευχαριστώ για όλη τη δουλειά σας Είδαμε σε προηγούμενες επισκέψεις με την αντιπροσωπεία Μερκοσούρ τι πρόοδος έχει επιτελεστεί. Είναι μια στατική συμφωνία αυτή και θέλουμε να πούμε ότι η κυβέρνηση της Παραγουάης, η τωρινή και οι προηγούμενες, έχουν υποστηρίξει την ε, επίτευξη μιας συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνία λοιπόν, όπως έλεγα, στατηγική, όχι μόνο από εμπορική σκοπιά, τα ξέρει και ο συνάδελφος εδώ καταλεπτός, αλλά και για άλλους πυλώνες συνεργασίας, ιδίω αυτόν του πολιτικού διαλόγου, που είναι πολύ σημαντικός, συνουσιώδης, για να υπάρξει σταθεροποίηση στις σχέσεις μεταξύ μας σχέσεις που δεν είναι μόνο οικονομικές, είναι και ιστορικές και πολιτικές. Έχει στατηγική σημασία και για τις δύο πλευρές η συμφωνία αυτή. Για μα υπάρχουν κάποιε προτεραιότητε που είναι ιδιαίτερα σημαντικέ. Τι έχουμε τονίσει με αφορμή τη συμφωνία και τι υπογραμμίζουμε εδώ και καιρό. Το είπε και ο Πρόεδρο στην παρέμβασή του. Η βιώσιμη ανάπτυξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι κλιματικέ αλλαγέ. Είναι θέματα επί των οποίων πρόκειται να εργαστούμε και περιμένουμε τους προσεχείς μήνες όπως θύμισε και ο Πρόεδρος αφού περάσουμε στη φάση χτενίσματος και μετάφρασης του κειμένου ε, μέσα στα επόμενα χρόνια να τα συζητήσουμε και στο Ευρωκοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια για τις λεπτομέρειες. Είναι σημαντικό η συζήτηση αυτή να συνοδευτεί από συγκεκριμένες προσπάθειες και αυτέ κινήσεις σε κάποια από τα θέματα αυτά τα οποία θύμισα και για μας πάνω απ' όλα μετράει να υπάρξει συνεργασία και για την ε, περιφερειακή συνεργασία των χωρών Μερκοσούρ μεταξύ τους, των τεσσάρων αυτών χωρών. Ελπίζουμε στο μέλλον να προσθεθεί και η Βενεζουέλα στις τέσσερις αυτές χώρες που για την ώρα έχει αναστείλει τις σχετικές συνομιλίες και τη συμμετοχή της στη συμφωνία. Ελπίζουμε λοιπόν να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την περιφερειακή συνεργασία και τις ιστορικές, πολιτικές, οικονομικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τεσσάρων χωρών του Μαρκοσούρ. Έχουμε εμπορική συμφωνία με τη Χιλή, τη Βολιβία, το Περού. Ε, Μα λείπουν οι χώρε του Μερκοσούρ για να έχουμε εμπορικέ συμφωνίε με τη Λατινική Αμερική. Όλε τι χώρε. Είναι σημαντικό λοιπόν για τι σχέσει μα με την Νότια Αμερική να προχωρήσουμε. Κύριε Υπουργέ, σα εύχομαι καλή επίσκεψη, καλού ε, διαλόγου αυτέ τι ημέρε τη Βρυξέλλη και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε και να είστε ένα από μία από τι κινητήριε δυνάμει και για τι υπόλοιπε χώρε του Μερκοσούρ και να προωθείτε τα θέματα τα οποία θέσαμε και εμεί ως προτεραιότητε. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Uh, Ευχαριστούμε κύριε Ντάντη. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Ρίβα για να μα ε, παρουσιάσει την άποψή του για τη συμφωνία αυτή. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, είναι τιμή για μένα που είμαι Υπουργό Εξωτερικών της Παραγουάη και έχω αναλάβει προσωρινά και την Προεδρία Μερκοσούρ, να βρίσκομαι εδώ και να μιλήσω μαζί σας ε, σε σχέση με την Συμφωνία Μερκοσούρ Ευρωπαϊκή Ένωση, που όπως είπε και ο Πρόεδρος, η αλήθεια είναι θα αποτελέσει και το αντικείμενο της παρουσίασής μου και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρόεδρο γι' αυτό. Είναι μια συμφωνία που κατέληξε στο ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα μετά από 20 χρόνια. Έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις, μερικές φορές συζητήσεις δύσκολες, αλλά το σημαντικό, και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω, είναι ότι η συμφωνία αυτή με την Ευρωπαϊκή Ένωση της Μερκοσούρ αποτελεί και το θρίαμβο της πελημερούς διάστασης απέναντι στην μονομερή διάσταση. Πρόκειται για δύο ε, περιφερειακούς ε, συνασπισμούς, ομάδες χωρών, ε, που έχουμε πολλά κοινά. Προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την ελεύθερη έκφραση, τον πολιτισμό. Υπάρχουν πάρα πολλές πτυχές που δείχνουν ότι μοιάζουν πολύ οι χώρε της μίας ομάδας με εκείνε τι άλλε χώρες. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσουμε στους πολίτες μας γιατί δεν υπήρξε συμφωνία ανάμεσα στη Μερκοσούρ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν ε, δεν προχωρήσουμε περισσότερο, μετά από ε, τόσα κοινά που έχουμε διαπιστώσει ότι έχουμε μεταξύ μας. Ε, οι επιχειρηματίες, οι Ευρωπαίοι, επεκτείνονται στη Λατινική Αμερική με αυτή τη συμφωνία. Και οι δύο πλευρές θα υποφεληθούν από τη συμφωνία αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το πλεονέκτημα να έχει πολύ μεταποίηση, υπηρεσίες και θα μπορέσει να ενισχύσει τα κέρδη της. Αλλά το κέρδος είναι και για τη Μερκοσούρ, γιατί πρόκειται για μια συμφωνία που τη χρειαζότανε με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς, ας πούμε, ως Παραγουάι, ούτε και άλλες χώρες, δεν είχαμε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα βασιστούμε λοιπόν σε αυτή τη συμφωνία και θα θέσουμε τις αναγκαίες βάσεις για μια οικονομική, εμπορική σχέση, πολιτική και συνεργασίας. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν βλέπουμε τη σχέση αυτή είναι ιδιαίτερα υποφελής και για τις δύο πλευρές. Πρόκειται για 88 δις και πρόκειται για πάρα πολλούς ε, κανόνες που θα αρχίσουν να ισχύουν τώρα και που θα μας επιτρέψουν να έχουμε ένα εμπόριο ελεγχόμενο και με ηρεμία να υποφεληθούμε από διάφορους κανόνες όπως για παράδειγμα στο τομέα του περιβάλλοντος ή στα εργασιακά, ώστε να προχωρήσουμε με τις σχέσεις μας αυτές. Επίσης, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τον κλάδο των υπηρεσιών, που επωφελείται οικονομικά. Υπάρχει Ε, για ένα ποσό 40 δις από τις υπηρεσίες. Επενδύει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Παραγουάη, για παράδειγμα. Και έτσι διαπιστώνουμε ότι αναπτύσσονται οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Μερκοσούρ. Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε και τους κανόνες που θα αρχίσουν να ισχύουν μεταξύ των δύο πλευρών. Εμείς περισσότερο από οτιδήποτε άλλο υπογραμμίζουμε ότι πρέπει να έχουμε μια συμφωνία με κανόνες. Αλλιώς να μην έχουμε συμφωνία. Γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε πολλού κλάδους σημαντικού για την περιοχή και επίσης όσοι Ευρωπαίοι που αποφάσισαν να επενδύσουν στις χώρες Μερκοσούρ και το έχουν κάνει εδώ και πολύ καιρό, θα μπορούν να βασιστούν σε μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απορρέουν από τις ίδιες τους τις χώρες. Έτσι νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολα τα πράγματα και με μεγαλύτερη τάξη, πιο συντεταγμένα. Οι χώρες Μερκοσούρα κάναν μεγάλη προσπάθεια για να καθορίσουν τους τομείς συνεργασίας και προκειμένου να δούνε πού προσφέρει ευκαιρίες η συμφωνία αυτή. Όπως το είπε και ο Ευρωβουλευτής Ντάντι, η Μερκοσούρ, οι χώρες Μερκοσούρ ήταν η μόνη ομάδα χωρών που δεν είχε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση από ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Άρα λοιπόν χρειαζόταν η συμφωνία αυτή πράγματι ξεκίνησε πριν από 21 χρόνια σε επίπεδο διαπραγμάτευσης δηλαδή. Το 1991 φτιάχτηκε η Μερκοσούρ και το πρώτο που έκαναν οι υπουργοί των χωρών Μερκοσούρ ήταν να έρθουν στις Βρυξέλλες και να δουλέψουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τους υπουργούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους τότε, των τότε 12 χωρών, γιατί θεωρήσαμε ότι υπάρχει κάποια αντιστοιχία ανάμεσα στις χώρες Μερκοσούρ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλαμε τεχνική ε, συνεργασία στον τομέα της Γεωργίας, για παράδειγμα, και το 1995 είχαμε και την πρώτη πολιτική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Το 1999 άρχισαν οι διαπραγματεύσεις και έτσι είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε εδώ αυτές τις εξελίξεις και την συμφωνία που υπάρχει μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μερκοσούρ σε πάρα πολλούς τομείς. Επαναλαμβάνω, η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα θρίαμβο της πολυμερούς διάστασης. Είναι πολύ σημαντικό να έχει η Μερκοσούρ συμφωνίες και με άλλες περιοχές του κόσμου με τις χώρες ΕΦΤΑ, και θα υπογραφεί αυτή η συμφωνία σύντομα. Επίσης, έχουμε προχωρήσει σημαντικά και σε συμφωνία με τον Καναδά, την Κορέα, τη Σιγκαπούρη. Όλα αυτά αποτελούν μία βάση για την Μερκοσούρ προκειμένου να τοποθετηθεί στον κόσμο εκτός Μερκοσούρ. Και πρέπει να σας πω και το εξής, πέρα από το ότι πρόκειται για συμφωνία μεταξύ κυβερνήσεων, Τώρα η συμφωνία αυτή Μερκοσούρ θα επεκταθεί περισσότερο ανεξαρτήτως κυβέρνησης, θα πρόκειται για συμφωνία κρατών και θα ενεργοποιηθούν έτσι διάφοροι πολιτικοί μηχανισμοί επίσης ε, στις χώρες Μερκοσούρ. Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, προστασία του περιβάλλοντος. Εγώ ξέρω για την ε, Παραγουάη έχουμε τον πρόεδρο Μάριο Άλντο Μπενίτεθ και το πρώτο που έκανε ήταν ότι πήγε στο Υπουργικό Συμβούλιο, στον Υπουργό Περιβάλλοντος, που ονομάστηκε Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, προκειμένου να κινητοποιηθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί, ώστε να έχουμε μία πολιτική περιβάλλοντος που να καταπολεμά την κλιματική αλλαγή στην Παραγουά. Η Παραγουά είναι μια χώρα που δεν ρηπαίνει σχεδόν καθόλου. Οι εκπομπές μας διοξιδίου του άνθρακα είναι περίπου ανύπαρκτες. Αυτό που κάνουμε λοιπόν εμείς είναι ότι προσπαθούμε να μειώσουμε την ρήπαση που προκαλείται από άλλες χώρες, όχι από μας. Θέλουμε βέβαια και κάποια πληρωμή για τα αποτελέσματα. Εξού και συνεργαζόμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε μέσω του Πράσινου Ταμείου να μπορέσουμε να έχουμε αρκετά κονδύλια για να συνεχίσουμε και να βελτιώνουμε τις συνθήκες περιβάλλοντος στην περίπτωση της Παραγουάη. Τώρα από εκεί και πέρα σας ευχαριστώ πολύ. Ό,τι ερωτήσεις έχετε είμαι στη διάθεσή σας. Και υπογραμμίζω ότι η συμφωνία αυτή σε πολιτικό, οικονομικό, εμπορικό επίπεδο αλλά και επίπεδο συνεργασίας μόνο ωφέλη θα φέρει και στις δύο περιοχές αυτές του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Έχουμε μερικά λεπτά για μια ανταλλαγή απόψεων, καθότι υπάρχουν αιτήματα και από τους ε, συναδέλφους. Ο κύριος Κάνιας, ε, που είναι εισηγητής της Επιτροπής ε, Ήτρε για τη Μερκοσούρ. Παρακαλώ, μείνετε στο ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πρέσβη και ευχαριστώ και τον Υπουργό. Χτες βρεθήκαμε και ανταλλάξαμε απόψεις και ήταν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ακούω αυτά που λέτε για το πόσο μεγάλη σημασία έχει η συμφωνία αυτή η Μερκοσούρ προκειμένου να υπάρξει πρόοδος όχι μόνο οικονομική, εμπορική αλλά και πολιτική και δημοκρατική κτλ. Η Παραγώ έχει κάνει πάρα πολλά βήματα και με μεγάλη επιτυχία παρόλο που ήταν δύσκολο μερικές φορές. Οπότε όντω αξίζει να ενισχυθούν οι προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στην Παραγουάη η Μερκοσούρ όντως αποτέλεσε μία όθηση για τα αποτελέσματα αυτά. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η συμφωνία πρέπει να επικυρωθεί τους επόμενους μήνες και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα αντιμετωπίσετε κάποιες δυσκολίες, προκαταλήψεις, έλλειψη γνώσεων, δυσπιστή κτλ. Οπότε επειδή εγώ είμαι ο εισηγητής για τη συμφωνία αυτή, θα ήθελα να μας εξηγήσετε ποια είναι τα ωφέλη για τους πολίτες, όχι μόνο τα μεγάλα ε, δεδομένα ότι θα εξάγουμε περισσότερο, θα έχουμε περισσότερα κέρδη κτλ. Όχι, για τους πολίτες της Παραγουάης. Τι σημασία έχει αυτή η ε, συμφωνία, ποιο είναι το φάσμα δηλαδή βελτιώσεων που θα διαπιστώσει ο πολίτης, περισσότερη δικαιοσύνη, περισσότερη προστασία του περιβάλλοντος, περισσότερη δημοκρατία, δεν ξέρω, για να ξέρουμε ότι δεν πρόκειται μόνο για το παρελθόν, αλλά πρόκειται και για ένα μέλλον κοινό που θα έχουν οι πολίτες της Μερκοσούρ με τους Ευρωπαίους πολίτες. Από το ΕΛΚΟ, κύριος Μιγιάν Μόν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Και ευχαριστώ για τα λόγια σας. Εγώ πολύ χαίρομαι που ολοκληρώθηκαν διαπραγματεύσεις πράγματι πάνω από 20 χρόνια. Τώρα πιστεύω ότι θα έχουμε μια συμφωνία από την οποία θα υποφεληθούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Είναι ιστορική σημασία, με τεράστια πρόοδο. Σίγουρα θα υπάρξει μια μεγάλη αγορά. Πέρα πάντω από ότι οι δυσκολίε μπορεί να αντιμετωπίσουν διάφοροι κλάδοι, η συμφωνία αυτή είναι ιστορικής σημασίας με πάρα πολλά ωφέλη για όλου. Τώρα, πολιτικά μιλώντα επειδή εδώ στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων περισσότερο για τα πολιτικά συζητάμε, και εδώ πιστεύω ότι είναι μια σωστή συμφωνία. Εγώ πάντα έλεγα ότι η Λατινική Αμερική και η Ευρώπη είμαστε από τη φύση μας σύμμαχοι. Έχουμε κοινέ αξίες, έχουμε κοινή χριστιανική κληρονομιά, πιστεύουμε στην πολυμερή διάσταση βασιζόμαστε σε κανόνες κλπ. κλπ. Συνεπώς, πιστεύω ότι έχουμε και κοινούς στόχους. Συνεπώς, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής, περιβάλλον κλπ. Δεν είναι μόνο δηλαδή οικονομικό το ζήτημα, αλλά είναι και πολιτικό. Θα ενισχύσει η συμφωνία αυτή τους δεσμούς που είναι φυσικοί μεταξύ μας. Τώρα, υποφελούμε από την παρουσία σας εδώ για να πω ότι και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα υπάρξουν κάποιες δυσκολίες, αλλά θα καταλήξουμε σε θετικό αποτέλεσμα, πιστεύω. Τέλος, θέλω να σας ρωτήσω, εσείς από τη δικιά σας οπτική γωνία της Μερκοσούρ, πώς βλέπετε τις πολιτικές αλλαγές στην περιοχή σα, στην Αργεντινή π.χ. ή την στήριξη στη συμφωνία αυτή κυβερνήσεων που μόλις ανέλαβαν στις χώρες σας. Ευχαριστώ κυρία Ρένα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστούμε για αυτή την εισήγηση. Ομολογώ ότι ε, αισθάνομαι πολύ άνετα γιατί αν δούμε την Παραγουάη και την Ουρουγουάη στο πλαίσιο της Μερκοσούρ, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα μπορούσε να υπάρξει συμφωνία και με τέτοιες χώρες. Ιδίως εφόσον ε, έχουμε όλο αυτό το πλήρες πλαίσιο της Μερκοσούρ, θεωρώ ότι ε, έχουμε εκατομμύρια ε, πολίτες, μια μεγάλη γεωγραφική έκταση, όμως ε, καμία σχέση με την ε, Βραζιλία και την Αργεντινή. Ακόμα και αν έχουμε ερωτήματα να θέσουμε για τη Μαρκοσούρ, περισσότερο θα μας απασχολήσει το θέμα της Βραζιλίας και της Αργεντινής, όχι των άλλων δύο χωρών. Ε, και εγώ από μια πολύ μικρή χώρα προέρχομαι, από το Βέλγιο, με 10 εκατομμύρια πολίτε, που χθε πήρε μια ξεκάθαρη θέση κατά τη ε, συμφωνία τη Μερκοσούρ. Στο ε, Κοινοβούλιο τη Βαλονία καταψήφισαν τη συμφωνία. Κάποιοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να πούν μια τόσο μικρή χώρα παίρνει μια τόσο ρηξικέλευτη απόφαση, αλλά θεωρώ ότι και εμεί προερχόμαστε από δύο μικρέ χώρε. Παρ' όλα αυτά έχουμε φωνή και μήνυμα. Σε ό,τι αφορά το Μερκοσούρ, ένα πρώτο ερώτημα για τη Γεωργία. Σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Γεωργία αντιμετωπίζει δυσκολίε. Η Μερκοσούρ θα βελτιώσει τα πράγματα στην Ευρώπη. Ένα ερώτημα είναι αυτό. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα τώρα. Σήμερα, σε ό,τι αφορά τη Βραζιλία πιο συγκεκριμένα, έχουμε υφαρπαγή ε, εδαφών που ουσιαστικά στερεί ε, τους αυτόχθονες πληθυσμού από ε, την γη τους. Τι μπορεί να κάνει ο Μερκοσούρ ως προς αυτό για το περιβάλλον είναι μια χώρα, η δική σα, η οποία δεν συμμετέχει στην Συμφωνία των Παρισίων. Μπορεί αυτή η χώρα να αποτελέσει εταίρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα του κλίματο που μα απασχολεί όλου, για την Βραζιλία εκεί πάλι. Υπάρχουν πολλά στοιχεία προβληματισμού σε σχέση με αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Άννα Καρατσίνη. Ε, ε, Καλώς ήρθατε. Κύριε Ρίβας, είναι πολύ καλό που έχουμε αυτή τη συζήτηση εδώ σήμερα για να δούμε ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ποιες είναι οι δικές σας θέσεις. Θα συνεχίσω στα αγγλικά, γιατί μου είναι δύσκολο, τα ισπανικά μου δεν είναι και τόσο καλά. Όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι απαιτείται μια στενότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών Μερκοσούρ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι ε, πολύ χρήσιμο ε, και αν δούμε το πολιτικό πλαίσιο της Συμφωνίας Μερκοσούρ είναι πολύ σημαντικό γιατί συχνά μιλούμε για το εμπορικό κομμάτι μόνο και ε, αφήνουμε κατά μέρο το πολιτικό που είναι πολύ σημαντικό. Κανένα δεν αντιτίθεται στη συνεργασία Τώρα, σε ό,τι αφορά το εμπορικό σκέλο τη συμφωνία, είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα και θέλω να επισημάνω μία σύνοψη τη συζήτηση που κάναμε στην Ολομέλεια λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Εμεί, όσο έπρασινοι, θέσαμε επιτάπητο στο ζήτημα. Κατά πόσο δηλαδή η συμφωνία Μαρικοσούρ συμβαδίζει και συνάδει με το Green Deal, που είναι είναι απαρχίδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την επόμενη πενταετία. Πώ δηλαδή η οικονομία μα θα γίνει φιλική προ το περιβάλλον. Πώς ε, θα προωθήσουμε την Πράσινη Συμφωνία. Εμεί και άλλοι συνάδελφοι έχουν σοβαρέ αμφιβολίες για το κατά πόσο η εμπορική αυτή συμφωνία συνάδει με το Green Deal. Γιατί αν δείτε τι γεωργικές εξαγωγέ που θα αυξηθούν, αυτό απαραίτητα θα οδηγήσει και σε αυξημένε εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Ε, εξίσου μα απασχολούν ε, και άλλα μη δεσμευτικά πρότυπα και κανόνες σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα για χώρα όπως η Βραζιλία που ανέφεραν και οι συνάδελφοι από τους σοσιαλιστές, υπάρχουν λοιπόν σημαντικά προβλήματα. Μιλώντας βέβαια με συναδέλφους από τις χώρες Μερκοσούρ, υπάρχουν σημαντικές ανησυχίες για την απώλεια θέσεων εργασίας, ε, για το κλίμα, καθώς θα εξάγουμε πολλά ε, προϊόντα, γαλακτοκομικά, κρέατα εφόσον αυτά τα προϊόντα τα έχουμε και εμείς και εσείς, γιατί να τα στέλνουμε από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη. Διακόπτει ο Πρόεδρος ε, να μιλήσουν και άλλοι συνάδελφοι. Ναι, μάλιστα, κλείνω. Ήθελα μόνο να πω κάτι τελευταίο. Είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν υπάρχει έλλειψη κανόνων. Έχουμε ήδη το πλαίσιο κανόνων του ΠΟΕ με βάση οποίου οποίους ε, πραγματοποιούμε τι συναλλαγέ μα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν ήδη κανόνε. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Βιλανουέβα, από την ΚΟΕ. Καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και για τόσα μας είπατε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Μερκοσούρ είπατε ότι ήταν οι μόνες χώρες, οι Μερκοσούρ, που δεν είχαν συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς ε, δεν ε, λέμε ότι δεν θέλουμε να υπάρχουν αυτές οι σχέσεις, λέμε ότι με αυτή την εμπορική συμφωνία δεν είμαστε τόσο πεπισμένοι. Κατά τη γνώμη μας, το μόνο που κάνει είναι ότι προωθεί ένα μοντέλο το οποίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας οδηγεί σε μια τραγική κατάσταση την Ήπεθρο, για παράδειγμα, με συνέπειες ε, στην κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για εμπορικές συμφωνίες όπου παράγουμε ένα μήλο το οποίο χιλιάδες χιλιόμετρα πιο μακριά καταναλώνεται, το τρώει κάποιος, έχοντας ε, δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλη ρήπανση για την μεταφορά. Υπάρχουν πολλές φωνές λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν βλέπουν τόσο το ωφέλη της συμφωνίας αυτής, πέρα από τα μεγάλα νούμερα που αφορούν καθαρά το εμπόριο, τι γίνεται με την βιωσιμότητα, με το μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία από τις συνέπειες στον πρωτογενή μας τομέα, στη γεωργία, στην κτηνοτροφία. Και θα ήθελα συγκεκριμένα να σας ρωτήσω το εξή. Φαίνεται ότι η Αργεντινή είπε ότι θα προχωρήσει σε μελέτη αντικτύπου για τη δικιά της οικονομία. Ξέρετε αν θα το κάνουν και άλλες χώρες ε, Μερκοσούρ και αν θα δημοσιευθούν τέτοιες μελέτες και μπορεί να επικυρωθεί μια τέτοια συμφωνία εάν μόνο δύο ή τρεις χώρες Μερκοσούρ την υποστηρίζουν. Η κυρία Γκονζάλης τώρα από τους σοσιαλιστές παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Ρίβας και κύριε Μαρικοαντώνιο. Για τη Συμφωνία Σύνδεσης, Μερκοσούρ. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι μιλάμε για μια συμφωνία σύνδεσης. Κάτι πολύ ευρύτερο από μια εμπορική συμφωνία. Και άρα συμπεριλαμβάνεται και ένα κεφάλαιο για πολιτικό διάλογο. Η δικιά μου πολιτική δύναμη και εγώ ίδια ε, πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλό να μπορούμε να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα πέρα από τόνους δημητριακών κρέατος και δεν ξέρω τι. Να συμπεριλάβουμε και αυτό ακριβώς κάνουμε και αυτό ίσως είναι που θα έπρεπε να ενισχύσουμε ό,τι έχει να κάνει με την συνεργασία για την ανάπτυξη, την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, περιβάλλον κλπ. Οπότε συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για το ότι τόσο η Παραγουάη όσο και οι άλλες χώρες μέλη της Μερκοσούρ είναι χώρες που έχουν κάνει καλά τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο για το περιβάλλον π.χ. και δεν θα πρέπει να τη συγκρίνουμε με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό να περάσει η συμφωνία αυτή, αλλά βέβαια όχι με οποιοδήποτε τρόπο. Μην βιαστούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που στο κάτω-κάτω 20 χρόνια χρειάστηκαν για να προχωρήσει στη διαπραγμάτευση. Μήπως θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερο για κάποια κεφάλαια, να τα δούμε λίγο περισσότερο σε βάθος και να δούμε πώς συνδέουμε αυτές τις δύο περιοχές του κόσμου που έχουν πάνω από 300 εκατομμύρια ε, ανθρώπους πληθυσμό. Χτες είχαμε τους αγρότες του Νότου που ήρθαν εδώ σε μια εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και λέγανε ότι πέρα από τις ζωοτροφές ε, που ταΐζουν τις, ε, τα ζώα μας εδώ στην Ευρώπη και μας έρχονται από εκεί, έχουμε και πάρα πολύ καλαμπόκι. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και καλό είναι να μιλάμε για όλα τα θέματα και μην ξεχνάμε ότι ναι, συμφωνία με την Μερκοσούρα, αλλά με περισσότερα δικαιώματα για τους εργαζόμενους, περισσότερα δικαιώματα για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και στη συνεργασία για την ανάπτυξη. Να δώσω το λόγο στον κύριο Ρίβα για να απαντήσω όσο δυνατόν περισσότερε ερωτήσει. Πολύ δύσκολο αυτό που σα αναθέτουμε. Πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω συνοπτικά κάπως να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Ναι, για την Παραγωγή είναι πολύ σημαντικό Από το 1989 ξεκίνησε τη δημοκρατική της διαδικασία Παραγουάη και είναι καλό να ανοίγει προς τον κόσμο Παραγουάη και ο κόσμος να ανοίγει τις πόρτες του στην Παραγουάη. Εξού και είχαμε τη συμφωνία συνεργασίας διμερός με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έφερε πολύ ωφέλη στην Παραγουάη. Πρώτα απ' όλα ε, από πλευράς δημοκρατίας. Δεύτερον, όσον αφορά την συνεργασία για την ανάπτυξη και ήταν και ένας δρόμος προς την Ευρώπη, κάτι το οποίο πάντα ήθελε η Παραγουάη. Στις περισσότερες φορές που ψηφίσαμε στην Παραγουάη είχαμε παρατηρητές των εκλογών από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Επίσης, πιστεύουμε ότι στις επόμενες εκλογές θα πρέπει να υπάρξει αυτή η συνέχεια και να έχουμε παρατηρητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία αυτή, Μερκοσούρ Ευρωπαϊκή Ένωση, θα διευκολύνει όχι μόνο τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά ε, θα μας βοηθήσει και πολιτικά. Μην ξεχνάμε ότι η συμφωνία αυτή έχει ένα πολύ σημαντικό πολιτικό περιεχόμενο συνεργασίας και θα μας προσφέρει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τις εξωτερικές απειλές δεν τις έχει μόνο η Ευρώπη και εμείς τις έχουμε στη δικιά μας περιοχή και είναι σημαντικό να μπορούμε να συνεργαζόμαστε και όσον αφορά την άμυνα και όσον αφορά την ασφάλεια και όλα όσα έχουν να κάνουν με την πολυμερή διάσταση προκειμένου να διατηρηθεί η συνεργασία μας και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις εξωτερικές απειλές που αντιμετωπίζει ο κόσμος σήμερα. Ε, με την Αργεντινή έχουμε συζητήσει και πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε σε επίπεδο Μερκοσούρ. Είναι μια κατάσταση που θα τη δούμε με την Αργεντινή αλλά και με τις άλλες δύο χώρες. Η Ουρουγουάη αναλαμβάνει από το Μάρτιο προκειμένου να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα όχι μόνο για τη Μερκοσούρ και κάθε μία από τις χώρες Μερκοσούρ αλλά και για ολόκληρη την περιοχή. Επίσης, όσο προχωράει η επικύρωση, κάθε χώρα της Μερκοσούρ, σύμφωνα με ε, το σχέδιό μας, θα έχει διμερός συζητήσεις. Για τη Γεωργία τώρα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι χώρες Μερκοσούρ βασίστηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιστορικά μιλώντας, και τηρούν όλους τους κανόνες, όλες τις απαιτήσει από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει πρώτον να διατηρήσουμε ε, το σύστημά μας εξαγωγών και θα ενισχυθεί το εμπόριο μεταξύ των δύο περιοχών. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια περιοχή του κόσμου όπου προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπου Ε, υπάρχει το Αμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου η κάθε χώρα αναλύει και παρουσιάζει τους νόμους και τους κανονισμούς που έχει όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ίδιο ισχύει και για τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Στην Παραγουάη, για παράδειγμα, έχουμε διάφορες συμφωνίες για την προστασία των ε, αυτόχθονων πληθυσμών και έχουμε πάει στο Διαμερικανικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για να επιστήσουμε την προσοχή σε αυτά που συμβαίνουν. Για το περιβάλλον, πάλι δουλεύουμε συντονισμένα με τη, στη Μερκοσούρ. Η προστασία του περιβάλλοντος μας είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το φυσικό περιβάλλον των χωρών Μερκοσούρ είναι μια περιοχή όπου έχουμε ηλεκτρική ενέργεια και αυτή χρησιμοποιούμε κυρίως που είναι καθαρή και την, ε, παράγουμε την ενέργεια αυτή από το νερό, είναι υδροηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχει συμφωνία για προστασία και αναδάσωση για την προστασία των δασών μας, δηλαδή επίσης και για τη μείωση της φτώχειας από το σχέδιο αυτό θα αποφεληθούν 17.000 οικογένειες της Παραγουάης. Δεν έχω πολύ χρόνο. Δεν ξέρω, θέλετε να έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστούμε που ήρθατε κύριε Ρίβας και μας συγχωρείτε που σας πιέζουμε τόσο πολύ για το χρόνο, αλλά έχουμε πολύ φορτωμένη μερισσία διάταξη και να με συγχωρούν και οι συνάδελφοι που τόσες φορές τους διέκοψα, αλλά τόσο χρόνο είχαμε για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Κύριε Υπουργέ, θα έχουμε πολλές ευκαιρίες για τους ερχόμενους μήνες και τα προσεχή χρόνια να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας αυτής. Δεν είναι ούτε πρώτη το τελευταία μα συνάντηση. Σίγουρα θα μας απασχολήσει πολύ και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Αν χαρά μας να σας αποδεχτούμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Και δεσμεύομαι όντω να ξανάρθω εδώ στις Βρυξέλλες. Είναι τιμή για μένα. Τον Ιούνιο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μας θα έχει επίσημη επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στις Βρυξέλλες. Και τώρα να περάσω τη θέση του Προέδρου που μοιάζει με θρόνο στον συνάδελφό μου David McAllister.